Yes, if you're ready, you can start. You may start, please. Μπορείτε να αρχίσετε, αν είσαστε έτοιμος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε την ε, δυνατότητα να υποβάλω την υποψηφιότητά μου ενώπιον της Επιτροπής σας. Θα κάνω την παρουσίασή μου σε τρεις γλώσσες. De Αυτό που έχει σημασία είναι η ανανέωση, ο ανανεωτισμός. Δηλαδή, βλέπουμε νέα, με καινούρια μάτια, τον ρόλο του Ευρωπαίου Ομπουτσμαν και θέλω να δώσω ε, απαντήσεις στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Ένα νέο χαρακτηριστικό είναι ότι είμαι επαγγελματίας του τομέα. Ήμουν, όπως ξέρετε, ομοσπονδιακός ομπουτσμαν στην χώρα μου, στο Βέλγιο, από το 1997 μέχρι το 2005. Τώρα είμαι καθηγητής στην Μπρουζ στο, στο Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό και προβάλλω έναν εναλλακτικό τρόπο ε, επίλυσης των διαφορών. Επίσης είμαι νομομαθής. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να προωθήσω το ρόλο του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή και αυτό το κάνω και ως νομομαθής. Δηλαδή το δίκαιο πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι το αντίστροφο για μένα είναι πολύ χρήσιμο και αναγκαίο για να γίνει κανείς διαμεσολαβητής, διότι σε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωτικό να είναι κανείς νομομοθής για να προβάλλει υποψηφιότητα συνηγόρου του πολίτη. Επίσης γνωρίζω τα ευρωπαϊκά όργανα και τους θεσμούς, καθώς και τα ευρωπαϊκά γραφεία στο Λουξεμβούργο, Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, ε, Κοπενχάγη, μέσα στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης ε, Συνεργασίας και έχω δημοσιεύσει άρθρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη λειτουργία της. Ένα άλλο ε, ατού, ας το πω έτσι, είναι ότι ομιλώ πέντε ευρωπαϊκές ε, γλώσσες και πιστεύω ότι έχει σημασία να σεβόμαστε την ταυτότητα του καθενός και τη γλώσσα του που είναι αναπόσπαστο στοιχείο της προσωπικότητάς του και αυτό που έχει, ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή. Η τελευταία πτυχή της υποψηφιότητάς μου είναι ότι πρόκειται για μία ε, διαγενειακή, ας το πω έτσι, υποψηφιότητα. Είμαι 49 χρονών, μεταξύ δύο γενεών δηλαδή, και μπορώ να αντιμετωπίσω νέες προκλήσεις και να εργαστώ για να επιλύσω ε, σημαντικά ζητήματα. Πρόκειται για μια ηλικία μεταξύ δύο γενεών δηλαδή. Και πιστεύω ότι μπορώ να επιλύσω πολλά χάσματα. Θεωρώ για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ότι θα πρέπει να διδραματίσει σημαντικούς ρόλους σε ό,τι αφορά τους στόχους της ενίσχυσης της δημοκρατικής εποπτείας στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μέσω της, του ρόλου κλειδί, αν θέλετε, του διαμεσολαβητή, επιτυγχάνεται και καλύτερος έλεγχος σε εθνικό επίπεδο και ως κοινοβουλευτικός διαμεσολαβητής σημαντικό είναι να συνδράμει κανείς στα εθνικά κοινοβούλια για τον εκδροματισμό της ε, Ένωσης. Το κοινοβούλιο είναι το όργανο με την μεγαλύτερη νομιμοποίηση στο ιστορικό των της Ένωσης. Για να προσδώσει και αυτό το χαρακτήρα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν τρεις βασικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να εισέλθουν στον πυρήνα των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς η αρχή της διαφάνειας θα πρέπει να καταστεί η διαφάνεια χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 1 της συνθήκης. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει διαφάνεια σε, όλες τις, ε, σε όλα τα θεσμικά όργανα, σε όλες τις υπηρεσίες της Ένωσης και θα πρέπει λοιπόν να καταστεί προτεραιότητα υπαριθμών 1 για τον διαμεσολαβητή. Η λογοδοσία επίσης αποτελεί το δεύτερο στοιχείο, το δεύτερο από τις βασικές αυτές αρχές σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο και η τρίτη αρχή, η οποία είναι πολύ σημαντική, είναι ο πολιτισμός της εξυπηρέτησης. Αυτή λοιπόν η αρχή θα πρέπει να αποτελεί μια θεμελιώδη προϋπόθεση και θα πρέπει να τεθεί στον πυρήνα των υπηρεσιών και θα πρέπει να αποτελεί την του κάθε υπαλλήλου της Ένωσης. Θεωρώ ότι θα πρέπει ένας άλλος στόχος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή να είναι η ενίσχυση των θεμελιδών δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά την χάρτα των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά την ε, καταπολέμηση των διακρίσεων, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των ε, αναπήρων, σε ό,τι αφορά ζητήματα αλληλεγγύησης και το καθεξής. Αυτά πιστεύω είναι θεμελιώδη ζητήματα. Ένα τέταρτο στοιχείο είναι ότι ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να αποτελεί πηγή μεταρρυθμίσεων να προτείνει μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Για να τεθεί, αν θέλετε, η διαδικασία μεταρρύθμισης αυτή πιο πολύ στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του πολίτη. Και μεταρρύθμιση για να τύχουν αναγνώρισης οι αρχές καλής διαχείρισης και να εφαρμοστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι ο διαμεσολαβητής μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ πολιτών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη σκληρή δουλειά για να πετύχω τους στόχους που ανέφερα ο Άνω, θεωρώ ότι θα μπορούσα να βοηθήσω προκειμένου να υπάρξει συμφιλίωση μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης να αυξηθεί και η ευαισθητοποίηση του Ευρωπαίου υπαλλήλου για τον ρόλο που διδραματίζει ως βιτρίνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να γίνουν δράσεις για να βελτιωθεί η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον πολίτη. Και τώρα θα περάσω στις συγκεκριμένες προτάσεις που θέλω να προτείνω. Καταρχάς, ε, οι συγκεκριμένες δράσεις και προτάσεις θα εστιαστούν στην καλύτερη ευρωπαϊκή διαχείριση. Καταρχάς, για να εποπτεύεται η πλήρης εφαρμογή της καλής διοικητικής συμπεριφοράς, όχι μόνο από τα τρία βασικά θεσμικά όργανα, αλλά από όλες τις υπηρεσίες της Ένωσης, ειδικά μετά από τη σχετική απόφαση τον Οκτώβριο του 2008. Ένα άλλο στοιχείο θα ήταν ε, η ανάπτυξη ενός κοινού κώδικα καλής ε, διοικητικής συμπεριφοράς. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω ότι θα χρειαζόταν ε, διαθεσμικός διάλογος που θα εμπλέξει όλες τις υπηρεσίες, όλα τα θεσμικά όργανα. Και επίσης θα ήθελα να οριστεί καλύτερα ο όρος της κακοδιαχείρισης για να συμπεριληφθούν πιο πολλές πτυχές από τη σήμερα. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι θα έπρεπε να διοριστεί και ένας ε, υπεύθυνο για τη διαφάνεια σε κάθε, ξεχωριστά σε κάθε ευρωπαϊκό όργανο και υπάρχει και μια εξαιρετική σχετική έκθεση του κυρίου Κάσμαν. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται η θέση αυτή. Τέλος, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Και φυσικά να πάει πολύ παραπέρα από την εφαρμογή αυτή. Κατά δεύτερον, η ανάγκη να, να αυξηθεί η σημασία και η ευαισθητοποίηση του κόσμου σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Και να σας δώσω κάποια αριθμητικά στοιχεία. Υπήρξε αύξηση των καταγγελιών μεταξύ 2003 και 2008 κατά 28,5%. Να δούμε πόσες από αυτές τις καταγγελίες ήταν παραδεκτές. Η αντίστοιχη αύξηση ήταν 15% και κατά κεφαλή η αύξηση αυτή είναι λιγότερο από 1% επειδή οι καταγγελίες, οι έρευνες, ε, μάλλον τελικά η αύξηση, η μείωση των ε, ερευνών ήταν 16,3%. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα πρέπει να διαφημίζουμε πιο πολύ τα δικαιώματα των πολιτών να αναφέρονται και να προσφεύγουν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα καλύτερη ενημέρωση, καλύτερη συνεργασία με τον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί αποτελεί το καλύτερο μέσο για την επαφή με τους πολίτες και θα ήθελα συνεχή συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια να δημιουργηθεί ένα αποκεντρωμένο δίκτυο απεσταλμένων του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή σε συνεργασία με τη μόνιμη την προσωπία της ε, Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής με τα διάφορα κέντρα ενημέρωση στα κράτη-μέλη που υφίστανται ήδη και τέλος θα ήθελα να προτείνω οι διοικητικέ αποφάσεις να αναφέρουν το δικαίωμα του πολίτη να προσφεύγει στον διαμεσολαβητή. Αλλά όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν μαζί με καλύτερη καθοδήγηση των πολιτών όταν ε, κάνουν καταγγελίες. Και θα ήθελα λοιπόν να υπάρχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα προκαταρτικών ερωτήσεων. Θα πρέπει να μειώσουμε σημαντικά τον αριθμό των μη παραδεκτών καταγγελιών, γιατί σήμερα ανέρχονται σε 85% του συνόλου των καταγγελιών και αυτό μας εμποδίζει στο έργο μας και θα ήθελα να δημιουργηθεί ένας διαδραστικός οδηγός, ο οποίος θα είναι ίδιος για όλα τα θεσμικά σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις σχετικές ιστοσελίδες. Μία τρίτη σειρά δράσεων θα εστιαζόταν στην εντατικοποίηση της συνεργασίας. Είναι πολύ σημαντικό το σκέλος αυτό. Συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των ε, Ευρωβουλευτών. Ξέρετε ότι το λιγότερο από 10% των καταγγελιών έχουν υποβληθεί από ευρωβουλευτές. Σε ό,τι αφορά δηλαδή καταγγελίες οι οποίες προέρχονται από την εκλογική περιφέρεια του κάθε βουλευτή. Αυτό καταδεικνύει ότι ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να βρει καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο για να υποβάλλονται τέτοιες καταγγελίες. Συνεργασία μεταξύ του διαμεσολαβητή και της Επιτροπής σας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε η συνεργασία ήταν πάντα εξαιρετική, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις και να αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμών και επίσης μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και άλλων επιτροπών, μεταξύ του Διαμεσολαβητή και των εθνικών ή περιφερειακών συνηγόρων και των σχετικών επιτροπών αναφοράς. Λειτουργεί το σύστημα, όχι όμως επαρκόξ. Το 2008 μόνο 8 νόμοι ξεκίνησαν από τέτοιες κοινέ δράσεις. 8 μόνο δεν αρκούν φυσικά αυτοί οι αριθμοί. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τις συνέργειες στο δίκτυο αυτό. Ζητώ επίσης μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ διαμεσολαβητή και των Εθνικών Επιτροπών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να εφαρμοστεί ο δοσμευτικός χάρτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τέλος μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για περιπτώσεις συνεχούς και επανελειμμένης κακοδιαχείρισης, όπου έχουν ε, εκδοθεί συστάσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Τέταρτη και τελευταία σειρά δράσεων και προτάσεων έχει να κάνει με τη βελτίωση των δράσεων του ίδιου του διαμεσολαβητή. Ο διαμεσολαβητής θεωρώ ότι θα πρέπει να αναθεωρήσει την σωστή χρήση του άρθρου 226 και 228 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες επί παραβάση, όπως τα γνωρίζετε. Πρόκειται για ένα βασικό στοιχείο της ε, καλύτερης ε, ρύθμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα πλαίσια της οποίας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και διαδικαστικά θέματα, αλλά και θέματα επί της ουσίας. Θα πρέπει επίσης να βελτιωθεί η διάρκεια των ερευνών. Έχει ήδη βελτιωθεί κατά μέσο όρο 13 μήνες διαρκεί μία έρευνα, αλλά θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει συστηματική παρακολούθηση των κρίσιμων παρατηρήσεων, των ε, κριτικών που γίνονται προκειμένου να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στα εθνικά στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε περιπτώσει κακοδιαχείρισης. Και τέλος, ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να προωθήσει την πιο απλοποιημένη διαδικασία, πιο απλοποιημένη διαδικασία σε αντιμετώπισης και τις πιο απλοποιημένες λύσεις για την εξέβρεση συνένεση. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ βασικό σε ό,τι αφορά την επίλυση των διαφόρων. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αν έχετε ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας. Ε, Ξεκινάει η συζήτηση. Δίνω το λόγο στην κυρία Γκρουνή. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας κύριε Μονέ μας δώσατε πάρα πολλά στοιχεία, αλλά θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για το, την επόμενη θητεία του Ευρωπαίου ε, Διαμεσολαβήτη. Ποιες είναι οι βελτιώσεις που προβλέπετε για το ρόλο του Διαμεσολαβήτη και εάν πιστεύετε ότι θα αλλάξει ο κανονισμός, η θέση του Διαμεσολαβήτη. Πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη τη συγκεκριμένη ευθύνη του διαμεσολαβητή όπως ορίζεται από τις συνθήκες και χωρίς να μιλήσω για συγκεκριμένα πρόσωπα, ποια είναι τα χάσματα ή τα κενά που διαβλέπετε στη θέση αυτή μέχρι τώρα. Πώς θα θέσετε σε εφαρμογή το σχέδιό σας, γιατί ίσως είναι δύσκολο να ε, καταφέρει κανείς τα πάντα πώς θα συνεργαστείτε με την Επιτροπή Αναφορών, αν μπορείτε να μας μιλήσετε συγκεκριμένα και πώς προβλέπετε τη συνεργασία σας με τα άλλα θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μποσινάρου. Ευχαριστώ. Κύριε Μονέ, η Επιτροπή Πέτη με ανησυχία ανέφερε ότι το 2008 ότι το 36% των προσφυγών σχετίζονται με την έλλειψη διαφάνειας και έλλειψη ε, πληροφόρησης ή μη χορήγηση πληροφοριών και εγγράφων. Πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτό έτσι ώστε να ε, οικοδομήσετε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ποια είναι η πρότασή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Άγκης. Ε, ε, Ευχαριστώ. Κύριε Μονέτ, θα ήθελα να σας υποβάλω μία σειρά σύντομων ερωτήσεων που σχετίζονται με όλα όσα μας παρουσιάσατε ανάμεσα στους στόχους σας, δηλαδή η βελτίωση της εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ύψης της σημασίας, διότι εργαζόμαστε για τον Ευρωπαίο πολίτη και όχι το αντίστροφο. Η πρώτη μου ερώτηση έχει ως εξής. Ποιες εγγυήσεις μπορείτε να μας παράσχετε έτσι ώστε να μην υπάρχει παραβίαση δικαιωμάτων έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης ισότητα δικαιωμάτων όλων των προσφευγόντων. Να μην υπάρχει πολίτης δεύτερης κατηγορίας για γεωγραφικούς λόγους ή για τη χώρα στην οποία ανήκει. Μιλήσατε στην αρχή της παρέμβασής σας για μία νέα ε, όθηση, όθηση σε σχέση με το χάσμα των γενεών θα μελετήσετε όλες τις ε, περιπτώσεις όπου υπάρχουν ε, υποψίες διαφθοράς, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για, τις υψηλότερα, για τα υψηλότερα κλιμάκια ενός κρατικού μηχανισμού. Όταν μιλάμε μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας, πολλές φορές έχουμε να κάνουμε με αντικρουόμενες, όχι αντικρουόμενες, αλλά θέσεις που βρίσκονται η μία στον αντίποδα της άλλης. Μιλάμε για καταπολέμηση τρομοκρατίας, για οργανωμένο έγκλημα και ούτω καθεξής. Δεν πρέπει να υπερβούμε ε, με ορισμένες οριοθετήσεις που έχουν γίνει. Θα ήθελα τη γνώμη σας ως προς το συσχετισμό μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας. Επίσης και μία άλλη ερώτηση. Με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας θα μπορούν να υπάρξουν και άλλες αναφορές σε σχέση με δημοψηφίσματα. Σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων μειονοτήτων που είναι συλλογικά δικαιώματα, όπως γίνεται τώρα στη Σλοβακία, όπου υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων της ε, ουγγρικής ε, μειονότητας. Πώς θα αντιμετωπίσετε τα θέματα αυτά, γιατί η ουγγρική μειονότητα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μητρική της ε, γλώσσα. Κύριε Παλιαδέλη. Ευχαριστώ πολύ Εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μωρέτ, για την πολύ δυναμική παρουσίαση ε, όσων πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν προκειμένου ο Ευρωπαίος Μεσολαβητής να ανταποκριθεί στο όραμα που έχετε εσείς δημιουργήσει για αυτόν. Μία πολύ απλή ερώτηση. Πώς σκέφτεστε να μειώσετε τη διάρκεια των ευρωπαϊκών των, των ερευνών που, έχουν σχέση με τον Ευρωπαίο Μεσολαβητή. Reduce the duration of the uh, European Ombudsman inquiries. Practically, meaning. Yeah? Ευχαριστώ. Χάρκιν, ευχαριστώ πρόεδρε. Και καλησπέρα σας κύριε Μονέτ. Σας ευχαριστούμε για την ε, πολύ εμπεριστατωμένη και πρακτική παρουσίαση που μας κάνατε. Έχω κάποιες ερωτήσεις που θέλω να θέσω. Σύντομες. Και θα ήθελα κυρίως να σας ζητήσω να μας δώσετε παραδείγματα για τα θέματα που θίξατε στην παρουσίασή σας. Μιλήσατε για το πώς θα περάσουμε από τα κλασικά νομικά ένομα δικαιώματα στις ένομες νομικές προκλήσεις. Τι ακριβώς εννοείτε. Θα μας δώσετε ένα παράδειγμα. Επίσης αναφέρατε στην επιχειρηματολογία σας τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του υπηρετικού, του ευρωπαϊκού και του αγγλοσεξονικού συστήματος, νομικού συστήματος και ότι υπάρχει ανάγκη φυσικά να γίνουν και τα δύο σεβαστά, αν θα θέλετε να αναπτύξετε το θέμα αυτό. Επίσης είπατε ότι ο νόμος πάντα θα πρέπει να είναι στην υπηρεσία του πολίτη. Έχετε κάτι συγκεκριμένο υπόψη σας κάποια συγκεκριμένη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς μπορούν καλύτερα να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του πολίτη. Τέταρτη ερώτηση. Μιλήσατε για κακοδιαχείριση και ότι θέλετε να διευρυνθεί ο ορισμός αυτός. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοούσατε, αν θα μπορούσατε να επαναλάβετε παρακαλώ. Και τέλος, μιλήσατε για την ανάγκη μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και της Επιτροπής Αναφορών σε ό,τι αφορά την ε, διερεύνηση των ίδιων θεμάτων. Έχετε κάτι συγκεκριμένο υπόψη σαν σας, αν θέλετε να μας δώσετε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Πολλά υπόσχονται αυτά που μας είπατε. Είπατε ότι θα βελτιώσετε την παρακολούθηση των διαδικασιών επί παραβάση και το είπατε αυτό και όσον αφορά τη διαδικασία και όσον αφορά το περιεχόμενο των δράσεων τη Επιτροπή στον τομέα αυτών. Μπορείτε να μα εξηγήσετε περαιτέρω πώ θα παρακολουθείτε τι αποφάσει τη Κομισιόν επί τη ουσία. Και επίσης είπατε ότι ελάχιστες φορές, ίσως ποτέ, οι, βουλευτές, οι ευρωβουλευτές δεν έχουν ε, ασκήσει το δικαίωμα τους να προσφύγουν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Πού σας λείπουμε, πού θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει καλύτερα τη δουλειά μας. Τι υποθέσεις θα έπρεπε να έχουμε υποβάλει στον διαμεσολαβητή, διότι αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Μας κατηγορείτε, μπορεί να έχετε πολύ σοβαρά πράγματα κατά νου που παραλείψαμε. Και είμαι πολύ περίεργη να ακούσω Πού δεν κάναμε σωστά τη δουλειά μας. Ο κύριος Σαλαβράκος. Αναφερθήκατε, κύριε Μωρέ, σε μια ισορροπία σχέσεων Όμπουσμαν και Επιτροπής Αναφορών. Και θα παρακαλούσα να μου πείτε, εάν βλέπετε κάπου θεσμικά να υπάρχουν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και ποιες είναι κατά την άποψή σας που δημιουργούν μια δυσλειτουργία στην άσκηση των καθηκόντων και των δικαιωμάτων του Όμπουσμαν. Ευχαριστώ. La parola di nuovo, Mr. Monet. Um, a lot of questions, Mrs. President. Πολλές ερωτήσεις, Πρόεδρε. Ελπίζω να μην ξεχάσω καμία. Κυρία Γκρούνη, σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που μου θέσατε. Με ρωτήσατε Ποιε είναι οι προτεραιότητες Ποια είναι μάλλον η προτεραιότητα την οποία ξεχωρίζω μεταξύ των όσων ανέφερα. Πολύ δύσκολο να ξεχωρίσω μία, γιατί φυσικά πολλά θέματα είναι κατεπήγοντα. Θεωρώ ότι αν θα έπρεπε να ξεχωρίσω μία προτεραιότητα θα ήταν το δικαίωμα των πολιτών να προσφεύγουν στον διαμεσολαβητή και νομίζω ότι το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να κατοχυρώνεται σωστά και αυτό θα αποτελούσε την κορυφαία προτεραιότητά μας γιατί η θέση του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή υπάρχει εδώ και 14 χρόνια και βλέπουμε όντως να αυξάνεται ο αριθμός των ε, καταγγελιών Κοιτώντα όμω τα αριθμητικά στοιχεία σε κάποιε ορισμένε χώρε βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση. Αλλά σε ό,τι αφορά το παραδεκτό των καταγγελιών, βλέπουμε ότι είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό αυτό. Γιατί δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, αλλά στο πεδίο αρμοδιότητα του Εθνικού Διαμεσολαβητή. οι πολίτες οι οποίοι έρχονται σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν μια πολύ μικρή ομάδα. Μπορεί τελικά να καταλήξουμε να έχουμε εκατομμύρια προσφυγές αν είναι υπερβολικά ευρύς ο ορισμός, αλλά είναι μικρός αριθμός των ε, προσφυγών για τις οποίες είναι τελικά αρμόδιο ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό επειδή και ο προϋπολογισμός ε, του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή επικρίνεται σε πολλές περιπτώσεις από τους Ευρωπαίους, από τους Ευρωβουλευτές. Μπορεί να θεωρήσει κανείς δικαίως ε, εκ πρώτης όψεως ότι ξοδεύονται πολλά χρήματα για να αντιμετωπιστεί μεγάλος αριθμός μη παραδεκτών προσφυγών. Τουλάχιστον στο Βέλγιο επικρατεί αυτή η άποψη. Θα πρέπει λοιπόν για πολλούς και διάφορους λόγους να τονίσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο σχετικά με το δικαίωμά του να αναφέρεται και να προσφεύγει στον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή. Ιδιαίτερα και με την ηλεκτρονική οδό για να διασφαλίσουμε ότι τελικά οι καταγγελίες που καταλήγουν σε εμά είναι οι καταγγελίες επί των οποίων μπορούμε να βοηθήσουμε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τροποποιηθεί το καταστατικό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Πριν από τέσσερα χρόνια ήμουνα υπέρ της αναθεώρησης αυτής για συγκεκριμένους λόγους, τρεις συγκεκριμένους λόγους, αλλά Δύο εξ αυτών έχουν πλέον αλλάξει. Θα ήθελα λοιπόν οι αλλαγές αυτές να συμπεριληφθούν και να εφαρμοστούν. Και το άρθρο 4.3 επιτρέπει στον διαμεσολαβητή να ε, έχει πρόσβαση στα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 9 του, στο, στην παράγραφο 9 του άρθρου 149 σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα απόρριτα έγγραφα. Πρόκειται για μια πολύ ωφέλιμη διάταξη η οποία δίνει εγγύηση στους ε, πολίτες ότι τα απόρριτα έγγραφα θα παραμείνουν απόρριτα. Là, précisément, αλλά όταν κάτι τέτοιο το λέει η διοίκηση, υπάρχει πάντα η υποψία της μεροληψίας. Όχι όμως όταν προβαίνει σε τέτοιες αποφάσεις ο διαμεσολαβητής. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ενισχύεται η εμπιστοσύνη του πολίτη. Άλλο ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω. Παρακολούθησα τη σχετική συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο αποφάνθηκε ότι δεν επρόκειτο για θετική δράση σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες, σε ό,τι αφορά την άμεση προσφυγή στο ΔΕΚ, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κακοδιαχείριση. Νομίζω ότι δικαίω αποφάσισε, όπω αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί με τη συνθήκη της Λισαβόνα, το Ευρωκοινοβούλιο έχει δικαίωμα προσφυγή στο ΔΕΚ και όντω με τον τρόπο αυτό υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης ε, της συνεργασίας του διαμεσολαβητή με το Κοινοβούλιο και της προσφυγής τους ε, στο ΔΕΚ. Για την ε, εφαρμογή του προγράμματος αυτού. Όντως είναι τεράστιο το έργο και έχω πολλά και διαφορετικά σχέδια για την εφαρμογή. Θα ήθελα να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργική και αποδοτική αυτή η θέση. Αλλά σε περίπτωση που με εκλέξετε θα είναι πενταετής η θητεία μου θα μπορώ να κάνω δύο πράγματα. Καταρχήν, να φροντίσω να υπάρχει καλή συνεργασία με τους ε, συναδέρφους μου, ώστε να τοποθετηθούν τα σωστά πρόσωπα στις σωστές θέσεις. Παρακολουθώ εδώ και 14 χρόνια τη δουλειά του διαμεσολαβητή και έχω εντυπωσιαστεί από τη δουλειά του πολύ καλά ειδικευμένου προσωπικού που έχει προσληφθεί. Δεν μπορεί να εφαρμόσει κανείς ένα τέτοιο σύστημα χωρίς να υπάρχει συνέργεια και βούληση για συνεργασία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα. Και πιστεύω εδώ ότι θα πρέπει να πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα. Θα πρέπει να προοδεύσουμε στο Βέλγιο, κανένας δεν ήθελε και κανένας δεν αναγνώρισε τον συνήγορο του πολίτη. Αναγνώριζε το ρόλο, αλλά ο διαμεσολαβητής θέλει να βοηθήσει, θέλει να βρει νέους τρόπους ώστε να αποφεληθούν όλες οι πλευρές και να εισαχθεί μια νέα φιλοσοφία στη συνεργασία. Καλή συνεργασία λοιπόν, καλό συντονισμό ανάμεσα στον διαμεσολαβητή, το προσωπικό και τα άλλα θεσμικά όργανα. Αυτό είναι στόχος μου. Και θα ήθελα να απαντήσω αργότερα στο θέμα όσον αφορά τη συνεργασία του διαμεσολαβητή με την Επιτροπή Μεταφορών, διότι τέθηκε επανειλημμένα η ερώτηση αυτή τρεις φορές. Και θα ήθελα να ε, πω ότι είναι πολύ σημαντική και η συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα για την εφαρμογή του ε, προγραμματός μου. Κύριε Ποστινάρο, είπαμε ότι το 75% όλων των ε, προσφυγών έχουν να κάνει με την έλλειψη διαφάνειας ε, και την άρνηση πρόσβασης στα έγγραφα. Αυτό είναι υπερβολικό. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό των εθνικών συνηγόρων του πολίτη. 36% λοιπόν είναι υπερβολικό ποσοστό. Είναι ανησυχητικό, δεν θα έλεγα ότι είναι ανησυχητικό, αλλά είναι σίγουρα σημάδι ότι ο διαμεσολαβητής, και αυτό έχει γίνει από τους δύο τελευταίους διαμεσολαβητές τα τελευταία 14 χρόνια, ε, θα πρέπει να ε, επικεντρωθεί η δουλειά του διαμεσολαβητή στη διαφάνεια. Και βέβαια βοηθιέται ο διαμεσολαβητής από τον ε, κανονισμό 1049. Αποτελεί μία από τις δυνατότητες προσφυγών για ανθρώπου που δεν έχουν τι πληροφορίε που θέλουν. Μπορούν είτε να προσφύγουν στο δικαστήριο είτε στον διαμεσολαβητή. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, όχι μόνο για τον διαμεσολαβητή ω ε, θεσμό, αλλά και για τους πολίτες ε, να γνωρίζουν ε, ότι ε, το δικαίωμα τους στην διαφάνεια γίνεται σεβαστό. Πώς μπορεί να αυξηθεί η διαφάνεια, πώς μπορεί να μειωθεί ο αριθμός προσφυγών για έλλειψη διαφάνειας προς τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Συνεργασία και γνώση είναι οι απαντήσεις. Συνεργασία με τα θεσμικά όργανα. Πρέπει να συνεχίσουμε να λέμε πόσο σημαντικό είναι δεν είναι τυχαίο ότι το άρθρο 1 της συνθήκης θέτει την διαφάνεια στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποθέτω ότι όπως και εγώ δεν έχετε εντυπωσιαστεί θετικά από το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στον Ευρωπαίο πολίτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έλλειψη διαφάνειας σίγουρα αποτελεί αιτία της έλλειψης εμπιστοσύνης. Πώς μπορούμε να ε, λύσουμε το πρόβλημα. Όλοι οι Ευρωπαίοι δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γνωρίζουν καλύτερα πόσο σημαντικό είναι όχι να υπηρετούν τα κοινοβούλια, τις κυβερνήσεις, τους πολίτες. Ο πολίτης έχει αξίωση στη διαφάνεια, σύμφωνα με τη συνθήκη. Οι υπάλληλοι λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα θέμα. Και εγώ ήμουν υπάλληλο Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η γνώση αυτή δεν είναι αρκετά διαδεδομένη. Έχει βελτιωθεί, αλλά υπάρχει υπάρχουν πολλά να γίνουν ακόμα. Και το δεύτερο στοιχείο είναι η συνεργασία. Πώς, όπως είπα στην κυρία Γκρίνη, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες. Μίλησα με έναν κύριο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεως. Όπως ξέρετε, έχουμε ένα μνημόνιο κατανόησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είπαμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό για, όλες, για όλους τους φορείς και για τον δικό του να έχουν τη διαφάνεια στον πυρήνα των καθημερινών τους εργασιών. Δεν τον γνώριζαν αυτό αρκετό, αρκετά. Γνώση λοιπόν και συνεργασία. Υπάρχουν νομικοί περιορισμοί, κάποιες ε, δεσμεύσεις ε, που θα πρέπει να εφαρμοστούν με την ευλογία των αρχών. Να απαντήσω στην κυρία Χάνκης. Συγγνώμη. Και εσείς με ρωτήσατε διάφορα πράγματα Δεν θα πρέπει να ανεβάσουμε το προφίλ του διαμεσολαβητή. Δεν θέλω να επικεντρωθώ υπερβολικά στον θεσμό του διαμεσολαβητή. Επικεντρώνομαι περισσότερα στο δικαίωμα προσφυγής του πολίτη στον διαμεσολαβητή. Αυτό θα πρέπει να γίνει πιο γνωστό. Με ρωτήσατε κάτι ενδιαφέρον. Μου θέσατε ένα κρίσιμο ερώτημα. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ισότητα των δικαιωμάτων. Αυτό αφορά και τον διαμεσολαβητή, όχι μόνο τον διαμεσολαβητή, αλλά και αυτόν. Να, εξασφαλίσει, να διασφαλίσει τον σεβασμό των δικαιωμάτων. Και όσον αφορά την ισότητα, εγώ θα πήγαινα πιο πέρα. Εγώ είμαι νομικό, όπω σα έχω πει. Έχω κάνει πολλέ δημοσιεύσει όσον αφορά το θέμα τη δικαιοσύνη. Δεν είναι ακριβώ η ίδια η έννοια της ε, δικαιοσύνης στο ε, αγγλοσαξονικό δίκαιο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο, στο δίκαιο των ε, χωρών της υπηρετικής Ευρώπης, υπάρχει έννοια της αλληλεγγύης. Αυτό με έχει καθοδηγήσει στη δουλειά μου, διότι στη δημόσια διοίκηση δεν μπορούμε να ασκούμε ένα καθήκον εάν δεν διασφαλίσουμε την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Δεν έχω αρκετό χρόνο να αναπτύξω την έννοια αυτήν που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι όμως ζωτικό στοιχείο σε μια δημόσια υπηρεσία όπου ο διαμεσολαβητής έχει να παίξει έναν ρόλο, μπορεί να βοηθήσει τη διοίκηση να γνωρίζει τα ζητήματα αυτά. Είναι αλήθεια, δεν έχω μιλήσει για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέχρι στιγμής. Και αυτό αποτελεί θέμα πυρηνικό θα έλεγα, θέμα πάρα πολύ βασικό για τον διαμεσολαβητή όπως είναι και για τον Όλαφ. Και επανέρχομαι στην ερώτηση της κυρίας Γκρινή. Χαίρομαι πάρα πολύ που το νέο καθεστώς του διαμεσολαβητή του δίνει το δικαίωμα να παραπέμπει υπάλληλο στον αρμόδιο φορέα όταν καταδεικνύεται ότι ε, υπάρχει διαφθορά. Η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιδεινωθεί από υποθέσεις διαφθοράς. Μπορεί να έχει κανείς χίλιους υπαλλήλους απόλυτα έντιμους, μία η υπόθεση διαφθοράς να έχει κανείς. Αυτό βγαίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι πολίτες το μαθαίνουν και η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδεινώνεται λόγω αυτής της μιας υπόθεσης. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε θέματα διαφθοράς. αλλά η αντιμετώπιση της, διαφθορής, της διαφθοράς γίνεται εκ των υστέρων. Η κατάρτιση γίνεται εκ των προτέρων. Θα πρέπει δηλαδή να διασφαλίσουμε οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι να είναι απόλυτα επαγγελματικοί στον τρόπο χειρισμού των θεμάτων τους. Ελευθερία και ασφάλεια. Είναι αλήθεια ότι το ένα δεν είναι ασύμβατο με το άλλο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ωστόσο, μερικές φορές μπορεί να υπάρχει μια αντίφαση. Μπορεί μπορεί στην ε, συνάντηση αυτή ελευθερίας και ασφάλειας να πρέπει να επαγρυπνεί ο διαμεσολαβητής ώστε να διασφαλίζει να υπάρχει από τη μία ασφάλεια, από την άλλη όμως να γίνεται σεβαστή η ελευθερία. Και είναι μεγάλη πρόκληση εδώ και αιώνες και θα παραμείνει η πρόκληση αυτή και τους επόμενους αιώνες. Η Ήπειρός μας έχει δημιουργήσει θεσμούς που επαγρυπνούν, που καυγίζουν ε, να το πούμε έτσι, στους ανθρώπους που δημιουργούν πολιτική εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην θυσιάσουν ε, την ε, ελευθερία στο βωμό της ασφάλειας. Και αναφερθήκατε και στις παραβιάσεις εις βάρος των μειονοτήτων. Καταλαβαίνω ότι ανησυχείτε, να το πούμε έτσι, όσον αφορά την, την ε, ξέρω ότι ανησυχείτε για τον, ε, την προστασία των δικαιωμάτων των ε, μειονοτήτων. Στη χώρα μου το Βέλγιο υπάρχουν τρεις μειονότητες. Πολύ με ενδιαφέρουν τα δικαιώματα των μειονοτήτων επί εννέα χρόνια. Φροντίζω φρόντιζα να γίνονται σεβαστές οι μειονότητες. Μπορεί όμως... Μπορεί όμως να, μην είναι πάντα φιλετικές οι μειονότητες, μπορεί να είναι γλωσσικές, ε, μπορεί να έχουν να κάνουν με το φύλλο. Αυτό αποτέλεσε σημαντικό θέμα για μένα επί 9 χρόνια και θα ήθελα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν έχω την ε, ευκαιρία, να συνεχίσω να δραστηριοποιούμε στον τομέα αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να επιταχύνεται, διότι έχουμε μείνει πίσω. Κυρία Παλιαδέλη, πώς μπορούμε να επιτυχύνουμε τη διαδικασία των ε, ερευνών. Χαίρομαι που θέσατε ερώτημα, διότι δεν θέλω απλώς να διασκορπίζω ωραίες ιδέες χωρίς να προτείνω τρόπους εφαρμογής. Αναγνωρίζω, όπως είπα εξ αρχής, ότι εγκρίθηκε το πλαίσιο ήδη και φτάνουμε στο 12ο μήνα, δηλαδή 12 μήνες είναι η μέση διάρκεια. Είμαστε στους 13, τώρα έχουμε μειώσει το χρόνο στους 12. Νομίζω ότι θα φτάσουμε στους 12 μήνες που είναι και η διάρκεια που αφορά τη διαδικασία του άρθρου 226 και 228. Ο ένας χρόνος είναι αποδεκτό και σε εθνικό επίπεδο, ε, αποδεκτή διάρκεια δηλαδή πώς μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό. Αυτό ήταν το τελευταίο σημείο που έθιξα χρησιμοποιώντας πολύ περισσότερο ε, λύσεις με βάση τη συνένεση και απλουστευμένες διαδικασίες. Αυτό το εφήρμοσα στο Βέλγιο, χρησιμοποιώντας το, τον πιο, τους πιο ευέλικτους χειρισμούς, κερδίζετε χρόνο, πολύ χρόνο, όπου εσείς και το προσωπικό σας στη συνέχεια μπορείτε να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στις έρευνες. Άρα θα πρέπει να εντοπίσουμε πώς ε, υπάρχει, ποιο είναι το πιο ευέλικτο πλαίσιο μεταχείρισης των προσφυγών έτσι ώστε να τις εντάξουμε στις πιο παραδοσιακές έρευνες. Έτσι έχω κάνει εγώ στη χώρα μου και έτσι νομίζω ότι μπορεί να γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κυρία Χάρκιν, Ε, κυρία Χάρκιν, όχι Όκεν, Χάρκιν, συγγνώμη γιατί κακοπρόφερα το όνομα. Μου υποβάλλετε μια σειρά ερωτήσεων. Δεν ξέρω κατά πόσο κατανόησα αυτό το πρώτο ερώτημα σε σχέση με τις ε, νέες προκλήσεις και τα παραδοσιακά δικαιώματα. Ως προς το δεύτερο ερώτημα, σύστημά σας η Ευρώπη βασίζεται στο common law, στο αγγλοσαξονικό σύστημα από την ε, άλλη πλευρά, το common law και το equity law, που είναι το αγγλοσαξονικό και το υπηρετικό δικαιοδοτικό σύστημα από την άλλη. Νομίζω ότι πρόκειται για συμπληρωματικά δικαιοδοτικά συστήματα. Όπως είπα και στην κυρία Χάνκης, στο Βέλγιο χρησιμοποίησα το equity law για να το εισαγάγω στο δικό μας νομικό σύστημα, στη δική μας χώρα. Και ήταν πολύ δύσκολο να πείσω το Κοινοβούλιο, τους ε, ορίζοντες τις πολιτικές και τους ακαδημαϊκούς ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι είναι μια αρχή που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για το νομικό μας σύστημα. Γι' αυτό πιστεύω στο συμπληρωματικό χαρακτήρα των δύο συστημάτων και νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο χώρο και στα δύο συστήματα στον τρόπο χειρισμού ε, των προσφύγων. Κάτι άλλο που θα ήθελα να αναπτύξω, αλλά δεν έχω χρόνο, είναι ότι στην Ευρώπη γνωρίσαμε τρεις ε, γενναίες ομπούτσμεν. δεκαετία του 70, η πρώτη γενναία στις σκανδιναβικές χώρες, μετά τις δικτατορίες σε πολλές χώρες και μετά την κατάρριψη του τείχους. Αυτές οι γενές ombudsman δημιούργησαν διαφορετικά χαρακτηριστικά και προτεραιότητες. Όλα τα συστήματα είναι χρήσιμα γιατί είναι συμπληρωματικά. Και αυτό είπα και εγώ. Γιατί θα πρέπει κανείς να είναι ombudsman για ολόκληρη την Ευρώπη μέσα στα πλαίσια των δύο συμπληρωματικών συστημάτων, συμπληρωματικών κατά τη γνώμη μου. Πώς ορίζω την κακοδίκηση. Όταν ο κύριος Σέντερμαν, ο πρώτος ομπουτσμαν, πρότεινε στο κοινοβούλιο Έχω την επιστολή που του είχα γράψει τότε, νομίζω το 96-97, όταν ε, του ζητήθηκε ο ορισμός της κακοδιαχείρισης, κακοδιοίκησης, είπε ότι θα πρέπει να καλύπτει την παραβίωση ενός δεσμευτικού νόμου ή αρχής. Και ήδη 14 χρόνια πριν διαφώνησε και το έγραψα όχι. Θα πρέπει να είναι ευρύτερος ο ορισμός. Η κακοδιοίκηση πρέπει να περιλαμβάνει τις παραβιάσεις του ήπιου νόμου μια αρχής, ακόμα και αν δεν είναι δεσμευτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κακοδιοίκηση σημαίνει παρανομία. Κακοδιοίκηση δεν σημαίνει υποχρεωτικά παρανομία. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούμε σε μια ευρύτερη ενιολογική βάση ως προς τον ορισμό. Τώρα θα ήθελα να, ερωτήσω, να απαντήσω σε ερωτήσεις που μου θέσατε ως προς συνεργασία μεταξύ Επιτροπής Αναφορών και Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Πιστεύω, επειδή παρακολούθησα την ιστορία αυτού του θεσμού, νομίζω ότι η συνεργασία μεταξύ Ombudsman, είδαμε τον κύριο Σέντερμαν, τον κύριο Διαμαντούρο, Στη συνέχεια η συνεργασία ήταν αγαστή με την Επιτροπή Αναφορών. Έχει βελτιωθεί, εν πάση περιπτώσει. Δεν επικρίνω τίποτα οι άλλες χώρες. Πιστεύω όμως ότι η συνεργασία είναι πολύ καλύτερη από ότι σε συνεργασία εθνικού επίπεδου. Ίσως ε, είναι ένα παράδειγμα προς από εθνικούς ε, συνηγόρους του πολίτη. Αυτό που είπα και η κυρία Παλιαδέλη είπε ακριβώς το ίδιο, είναι ότι για, σε θέματα επικάλυψης μεταξύ Ombudsman και Επιτροπής Αναφορών θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε περισσότερο για να μην έχουμε την, το διπλό φόρτο. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε ένα και περισσότερο να βρούμε ζητήματα ή προσφυγές όπου οι αναφορές αφορούν ε, μία συλλογική προσφυγή όπου ο Ομπούτσμεν ήταν δραστήριος και ίσως θα πρέπει να έχουμε περισσότερες ανταλλαγές πληροφοριών και επικοινωνία γενικά όταν εργαζόμαστε σε παρόμοια ζητήματα. Τώρα, κυρία Άουκεν, κυρία Αουκεν, μου υποβάλλατε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα νομικής υφής. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής μπορεί ή δικαιούται, ας το πούμε έτσι, να αποτιμήσει τον τρόπο που έχει χρησιμοποιήσει η Επιτροπή τα άρθρα 226 και 228, η χρήση τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπα ότι σε διαδικαστικά αλλά και σε θέματα ουσίας μπορούμε να κρίνουμε την χρήση, την κατάχρηση, την έλλειψη χρήσης αυτών των αρμοδιοτήτων και εξουσιών. Δεν λέω ότι ο ομπουτσμαν θα πρέπει να ελέγχει κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί αυτές τις δικαιοδοσίες του 226-228 το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ευρωπαίου Ομπουτσμαν και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δύο αυτά άρθρα ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διακριτική ευχέρεια χρήσης ημί του 226 και η διακριτική αυτή ευχέρεια μπορεί να επικριθεί, αλλά έχει ε, εγκριθεί από το ΔΕΚ, άρα δεν τίθεται εν κινδύνο. Άρα λέω ότι ο Ομπούτσμαν ήδη λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Αν διαβάσετε την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, βλέπετε ότι έτσι κινείται σε διαδικαστικά ζητήματα ή σε θέματα ουσίας για την εφαρμογή του 226. Ο Ombudsman μπορεί να ορίσει ότι η Επιτροπή δεν έκανε λογική χρήση του 226. Και τώρα στρέφουμε σε μια βασική αρχή που έχει αναπτυχθεί στο Βέλγιο, το θέμα του ευλόγου. Δηλαδή, κατά πόσο ένας φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει μια εξουσία και δεν μπορεί να την ε, ε, χρησιμοποιήσει εφόλους της ύλης. Δηλαδή, η διακριτική ευχέρεια δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά. Και αυτό αφορά διάφορα δικαστικά και δικαιοδοτικά όργανα. Δηλαδή, η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες της, αλλά με βάση μια ορθολογική χρήση όπως ισχύει και στην περίπτωση του διαμεσολαβητή, ο οποίος ξέρει ή θα πρέπει να γνωρίζει κατά πόσο το 226 ή 228 έχουν χρησιμοποιηθεί εύλογα. Δηλαδή, κατά πόσο έχουν χρησιμοποιηθεί ορθολογικά αυτά τα δύο άρθρα ή έχουν ε, ή, ή, έχουν, ε, έχει γίνει κακή χρήση. Ο κύριος Σαλαβράκος έχει φύγει, αλλά θα το απαντήσω. Είπα ότι δεν υπάρχει καμία ένταση μεταξύ της ε, δικής σας Επιτροπής και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή εδώ και 14 χρόνια αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να χτίσουμε μια στενότερη συνεργασία. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι αρχίζει η διαδικασία του Catch the Eye. Εντάχει μόνο ένα αίτημα έχω από την κυρία Χάπινγκ και θα της δώσω ένα λεπτό καθώς και ένα λεπτό για την απάντηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μιλάω Ολλανδικά γιατί και ο μιλητή μα μιλάει τόσο καλά ολλανδικά. Ακούγοντα λοιπόν το πρόγραμμά του μου φαίνεται τόσο φιλόδοξο όσο και του Ομπάμα. Πώς θα γίνει όμω αυτό, γιατί βρίσκεται σε μία απομόνωση στο Στρασβούργο. Εγώ εργάστηκα στο γραφείο του Επιτρόπου Κάλλα και ήμουν ο αντίθετος πόλος, αν θέλετε, του Ευρωπαίου Μεσολαβητή στο γραφείο αυτό και συχνά αναζητήσαμε φιλικές λύσεις. Συμφωνούσαμε τον ε, διαμεσολαβητή, αλλά η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας είπαν ότι «Α, όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται για τον τάδε ή δίνα λόγο» και υπήρχε μια έντονη, αν θέλετε, ε, προάσπιση της, των δικαιωμάτων του διαμεσολαβητή. Ήταν αρκετά άκαμπτη η στάση του. Σας ρωτώ λοιπόν πώς θεωρείτε ότι θα διαμορφωθεί ο ρόλος σας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γιατί είπατε ότι θέλετε να δραματίσετε ιδιαίτερα ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση και ότι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες τα δικαιώματά τους. Πώς θεωρείτε λοιπόν ότι τα δικαιώματα αυτά μπορείτε να τα διαφημίσετε στον τύπο. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι αν εκλεγείτε κάθε επιτυχία σε ό,τι αφορά την μεταρρυθμιστική σας αυτή η ατζέντα που θυμίζει ο Ομπάμα. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η ερώτησή μου ταιριάζει πολύ με αυτά που είπε ο προλαλή σα. Όταν ακουστεί, όταν οι πολίτες της Ευρώπης έχουν την εντύπωση, λάβουν την εντύπωση ότι ο διαμεσολαβητής μπορεί να κινήσει πολλά, τότε και οι προσφυγές θα αυξηθούν. Αν υπάρχει εντύπωση ότι δεν έχει κανένα νόημα, τότε δεν προσέγγει κανείς το διαμεσολαβητή. Πολύ ωραία ακούγεται και το υπογράμμισα ότι το πιο σημαντικό είναι να μην διαρκεί πολύ η προσφυγή. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι Τι θα πρέπει νομοθετικά να αλλάξει για να αυξηθεί η βελτίωση και χρειάζεστε τη βοήθεια του Κοινοβουλίου. Θέλουμε να πολεμήσουμε σε όλα τα μέτωπα και εμείς έχουμε το στόχο τις αναφορές να τις επεξεργαζόμαστε γρήγορα. Διότι ο πολίτης έχει δικαίωμα σε μια απάντηση και μάλιστα δικαίωμα σε απάντηση μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα. Τι πρέπει να αλλάξει, αυτό είναι το, το ερώτημά μου. Κύριε Επίνγκ, σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή που μου θέσατε. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικά φιλόδοξο το πρόγραμμά μου. Δεν ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι κανείς φιλόδοξος σε μια τέτοια θέση. Όντω είπα ότι ασχολούμαι εδώ και χρόνια στο πλαίσιο διαφόρων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέρω πόσο δυνατά μπορεί να είναι τα θεσμικά αυτά όργανα για την υπονόμευση μεταρρυθμίσεων. Όντως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ιδιαίτερα, παρουσιάζονται κατά καιρούς ε, παραδείγματα θεσμικά όργανα, υπάλληλοι οι οποίοι δεν είναι υπέρ των αλλαγών. Αυτό όντως αληθεύει. Αλλά αυτό αποτελεί και τμήμα, αν θέλετε, της καθημερινότητας των θεσμικών οργάνων και σε εθνικό επίπεδο είναι καθημερινό φαινόμενο ότι ο μεσολαβητής, ο συνήγορος του πολίτη, να ζητά διαρκώς αλλαγές, να ζητά διαρκώς ε, πιο πολύ διαφάνεια, πιο πολύ ανοιχτό χαρακτήρα και επί εννέα χρόνια ασχολούμαι με τέτοια ζητήματα. Ασφαλώς και τα πράγματα δεν γίνονται σε μία νύχτα. Και έμαθα να είμαι υπομονετικός αλλά και επίμονος. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα να επιτυχάνονται οι στόχοι μας. Αυτά δεν συμβαίνουν σε μία νύχτα, όπως είπα. Μου θέσατε και μια δεύτερη ερώτηση για το πώς θα προβάλλω το έργο μου, το έργο των συνεργατών μου στον τύπο, στο ΜΜΕ. Να χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα διάφορα χώρα, διάφορες χώρες. Τη Γαλλία, το Βέλγιο και το καθεξής όπου υπάρχουν ιδιαίτερες συμφωνίες με τον τύπο για να γνωρίσουν καλύτερα τα μέσα τη λειτουργία των θεσμικών αυτών ε, θέσεων. Δεν, είναι, δεν μιλάω απαραίτητα για συνέντευξης τύπους, τύπου, αλλά γενικά δράσεις για την προώθηση της ε, ευκρίνειας, αν θέλετε, του έργου του κάθε θεσμού. Δεν έχω πολύ χρόνο να απαντήσω στον επόμενο ομιλητή, αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να γεννηθεί μια ελπίδα στον κάθε πολίτη αν δεν γίνεται σεβαστή η ελπίδα αυτή. Συμφωνώ απόλυτα και Το έχω ζήσει, το έχουμε δει στο Βέλγιο, γιατί κάνει δεν είναι τέλειος. Όντως αληθεύει αυτό. Γι' αυτό λοιπόν και είπα ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε. για να γίνει πιο γνωστό το δικαίωμα του πολίτη να αποτανθεί στον διαμεσολαβητή και να αναπτυχθούν σχετικά προγράμματα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες δεν προσφεύγουν στο διαμεσολαβητή για θέματα τα οποία δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους. Δεν μπορούμε να κάνουμε το ένα χωρίς το άλλο. Θα ήταν πραγματικά τρομακτικό. Θα πρέπει να υπάρχει η σωστή συνεργασία στο επίπεδο αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Μονέτ. Έληξε η ακρόαση. Σας χαιρετούμε. Έχουμε λίγα λεπτά για να κλείσουμε με τις εργασίες μας. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή δεν έχει ούτε καθήκον ούτε εξουσία να αποφασίσει ή να ε, εκφράσει απόψεις μετά από αυτό το μαραθώνιο μπορούμε απλώς να διαβάσουμε στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου τα πρακτικά αυτών των ακροάσεων με όλες τις παρεμβάσεις και τις επεξηγήσεις ως προς τις τρεις αυτές ακροάσεις ε, των τριών υποψηφίων. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις ή υποδείξεις, Θεωρώ ότι μπορούμε να κλείσουμε τη συνεδρίαση.